Okay, friends. Uh, first... Καλημέρα σας. Να δώσουμε παρακαλώ στους διευμηνεί την δυνατότητα να μας διαβάσουν ένα πολύ μικρό κείμενο. Η διευμηνία σας ενημερώνει ότι είναι η 37η ημέρα σήμερα ε, διαμαρτυριών λόγω της άτεγκτης στάσης της διοίκησης στα πλαίσια του καθορισμού των νέων συνθήκων εργασίας και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θα μπορέσουμε να δεχθούμε οποιαδήποτε υπέρβαση ωραρίου. Ευχαριστώ. Okay, friends. Then Οπότε ας περάσουμε στην ψηφοφορία για το θέμα της προφορικής ε, ερώτησης προς το Συμβούλιο. Πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου για ε, κοινωνική προστασία των εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων. Άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται πανψηφί με 47 ψήφους. Θα ψηφίσουμε και την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρχεται η ψηφοφορία. Έτοιμα ερώτηση για προφορική απάντηση. Ψηφίσατε όλοι τέλο ψηφοφορία και εδώ παμψηφί με 49 ψήφους εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ θερμότατα και περνάμε στον κανονικό κατάλογο ψηφοφορία τη έκθεση για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωής για τους γονεί και τους φροντιστέ. Τροπολογία 263. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 28. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία μη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 264. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 265. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 266 καταπίπτει. Πάμε στην 267. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές απορρίπτεται. 268. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές απορρίπτεται. 269 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 20. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 21. Στην τέταρτη σελίδα του καταλόγου. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην πέμπτη σελίδα του καταλόγου ψηφοφορίας και στην τροπολογία, μάλλον στην έκτη σελίδα του καταλόγου ψηφοφορίας, στη συμβαστική τροπολογία 22. Πολύ σημαντικό θέμα. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία H. Ποιος είναι υπέρ? κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 23. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 24. 24. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 35 μαζί με την 340 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 339, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 341, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 342 και 343 και 344 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 345. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αλλά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε για την 345. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 26 ψήφι υπέρ. 348 καταπίπτει. Πάμε στην συμβαστική τροπολογία 25. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 361. Μαζί με τη Γιούρη 32. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Εναλλακτική τροπολογία 26α. Συμβαστική ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την εναλλακτική συμβαστική τροπολογία 26α. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας υπεράριθμος από τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές. Εντάξει, τώρα τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με 23 ψήφους κατά. Συμβαστική τροπολογία 26. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 384. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απόρι ηλεκτρονικός έλεγχος μάλλον για την 384. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία και απορρίπτεται 26 ψήφοι κατά. ΦΑΜ 39. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 388. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 389. Ποιος είναι υπέρ. Ή μάλλον καταπίπτει αυτή. Νομίζουμε τουλάχιστον ότι καταπίπτει 389. Όχι, τελικά πρέπει να ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 393. Ποιος είναι υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. 300

391. The second part. The second part. Second part. So if the first part, is false, and the second part is compatible, so it has to be Okay, we vote on the second part of 391. Δεύτερο τμήμα του 391. Άρχεται η ψηφοφορία. Μάλλον ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 396 καταπίπτει, 397 το ίδιο. Συμβαστική νη. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 27. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 414 τροπολογία. 414. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 414 έρχεται η ψηφοφορία. Ένας υπεράριθμος ε, σοσιαλιστής. Απορρίπτεται. 30 ψήφοι Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 32. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία I. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 424. ή μάλλον δεν χρειάζεται. Πάμε κατευθείαν στη συμβαστική τροπολογία 28. Ποιο είναι υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 430. Ποιο είναι υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 29. ποιο είναι υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 30. Ποιο είναι υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β. ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 39. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 31. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 466. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 469. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 457 έχει καταπέσει. Γιατί η συμβαστική 27 έχει εγκριθεί. Φαίνεται στον κατάλογο ψηφοφορίες. Άμα θέλει το συζητάμε αργότερα, αλλά έχει καταπέσει, ε, δεν υπάρχει αφιβολία. Συμβαστική 33, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 491. Τη βρήκατε. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 491. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 37 ψήφοι κατά. 492. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 494. Ή μάλλον πρώτα 492. Ψηφίσατε. Απορρίπτεται με 39 ψήφους κατά. «494. Προφορική τροπολογία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών». Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 494. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 25 ψήφοι υπέρ. Τροπολογία 495. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία J. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 503. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ ή μάλλον καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Οπότε πάμε στη συμβαστική τροπολογία 34. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 528. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 528. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται με 27 ψήφους. 529. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 529. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 28 ψήφους κατά. Τροπολογία 530 καταπίπτει. 530 μάλλον, γιατί δεν εγκρίθηκε 529, κατά αποχές απορρίπτεται. 531, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 35, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 της Επιτροπής Γυναικών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 545 καταπίπτει. Πάμε στην 546 προφορική των σοσιαλιστών. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 548. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 548 548 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ Σχεδόν οριακή διαφορά. Συμβαστική τροπολογία 36. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Κ. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 567. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 567. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 32 ψήφους κατά. Τροπολογία 571. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται. 572. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 573. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 578. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 577. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 574. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 574. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 39 ψήφους κατά. Τροπολογία 575. Ή μάλλον 500... Όχι, 575. 575. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 575. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is now closed. Τέλος ψηφοφορίας. Οριακά, με μία ψηφοδιαφορά απορρίπτεται. Τροπολογία 576. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ευχαρίστως. Άρχεται η ψηφοφορία για την 576. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με 33 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 580. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 579. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 581. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία L. Ποιο είναι υπέρ. Κατά απόχε. εγκρίνεται. Τροπολο... Συμβαστική τροπολογία 40. Ποιο είναι υπέρ. Κατά απόχε, εγκρίνεται. Τροπολογία 588. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχο για την 588. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 37. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 601. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 602 μαζί με την 603. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία 38. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 39. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 619. Ποιος είναι μαζί με την 620. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 621 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Απορρίπτεται. 622. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 622. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. ...623. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, 624 απορρίπτεται. 625 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 626 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 30 ψήφους κατά. Τροπολογία 628. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία για την 628. Τέλος ψηφοφορίας. Με 31 ψήφους κατά απορρίπτεται. Γιούρι 50, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη Γιούρι 50. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is soon Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 35 ψήφους. Τροπολογία 629. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 629, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 630 μαζί με την ε, τροπολογία 55 της Επιτροπής Γυναικών. Υπέρ κατά αποχές νομίζω πρέπει να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 29 ψήφους κατά. Τροπολογία 627 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 631 μαζί με την 51 της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 631 και την 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 30 ψήφοι κατά. Πάμε στην τροπολογία 632. Είναι προφορική τροπολογία από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Εντάξει, ας το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία. Πέρας και εγκρίνεται με 37 ψήφους. Πάμε στην ε, τροπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 633. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Εντάξει, να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 633 ηλεκτρονικά. πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με τρεις ψήφους. Πάμε τώρα Στη συμβιβαστική 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 649 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 650 51 συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 652 υπέρ καταπίπτει. 653 με την 6... Α, όχι, καταπίπτει και αυτή. Πάμε στην 58 της Επιτροπής Γυναικών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 669 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 670 μαζί με την 671 και την 60 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο άρθρο 19. Τροπολογία 676 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 20. Παράγραφος 1 και υποπαράγραφος 1. Τροπολογία 677. 677 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 678 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε να ψηφίσουμε την 679 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνουμε ηλεκτρονικά, ε, ναι, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 679 πέρας ψηφοφορίας Τι έγινε. Απορρίπτεται. Τι έγινε. Αλλάξατε στρατόπεδο κάποιοι. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην Γιούρι 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά την ε, τροπολογία 28. Πέρας ψηφοφορίας Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Ακαταπίπτει 29. Συμβιβαστική 2 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τσεροπολογία 35 μαζί με την 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά πάμε στην συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 43. Όχι, 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε τη 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται με 31 ψήφους. Τροπολογία 45 καταπίπτει. Ψηφίζουμε τη 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 53 μαζί με την 54 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 των Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά πάμε στην συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία αυτή καταπίπτει. Τροπολογία 83. Υπέρ. Κατά. Να την ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 83. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με τρεις ψήφους διαφορά. Γιούρι 11. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, 88 συγγνώμη, κατά αποχές εγκρίνεται. 9. μαζί με την 94, 9 της Επιτροπής Γυναικών, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 91 υπέρ, κατά αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 91. Πέρας ψηφοφορία. εγκρίνεται με 43 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 86 υπέρ. Κατά αποχέ, απορρίπτεται 92 υπέρ. Κατά αποχέ, απορρίπτεται 93 υπέρ. Κατά Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 93. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 32 ψήφους υπέρ. Υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε στην 95 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Γιούρι 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 97 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γιούρι 14, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 99, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 100, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η Γιούρι 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 17 της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γιούρ 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά πάμε στην τροπολογία 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 11 της Επιτροπής Γυναικών. Πέρας απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Amendment 153, yes. 153 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά πάμε στη συμβαστική 12. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 178. Όχι, κατά καταπίπτει. Άρα πάμε στη συμβιβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 181. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά πάμε στην τροπολογία 197 καταπίπτει. Πάμε στη συμβιβαστική 15 άρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 200. Μαζί με την 177. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν την τροπολογία 200 μαζί με την 177 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και όντως απορρίπτονται με μία ψήφο διαφορά. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές αγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 214. Ο, καταπίπτη. Άρα πάμε στη συμβαστική 17. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.16. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Α, να το ελέγξουμε. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 216. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. Συμβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18. Υπέρ. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική 18. Πέρας. Εγκρίνεται με 40 ψήφους. Υπέρ και 12 κατά. Πάμε στη συμβαστική Ι. E. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά πάμε στην 2.39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.40 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.42 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά πάμε στην τροπολογία 26, όχι, η τροπολογία 26 καταπίπτει. Πάμε στην 246, υπέρ,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 Πάμε στη 248 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 259. Καταπίπτει. Πάμε στο δεύτερο τμήμα της 259. Υπέρ κατά να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της 259. Πέρας πληροφορίας και απορρίπτεται με 32 ψήφους. Πάμε στην 261. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εντάξει, ελέγχουμε την 261 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία. Όχι. Τελική ψηφοφορία λοιπόν. Ε, το ΕΝΕΦ e θέλει να κάνει μια δήλωση μειοψηφίας Μήπω μπορούμε γραπτός να την έχουμε παρακαλώ μέσω της γραπτής διαδικασίας ευχαριστώ άρα ψηφίζουμε συνολικά την γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται με 34 ψήφου υπέρ, 14 ψήφου κατά και 4 αποχέ. Καλώ λοιπόν θα ψηφίσουμε τώρα για την εντολή. So the vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία για την εντολή. Πρέπει να υπάρξει φυσικά πλειοψηφία. Άνω των 28 θα πρέπει να υπερψηφίσουν πέρα της ψηφοφορίας. 37 υπέρ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα ξεκινήσουμε τις διοργανικές διαπραγματεύσεις.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

Όσοι παρακαλώ εγκαταλείπετε την αίθουσα να το κάνετε πάρα πολύ γρήγορα. Το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη θα ξεκινήσουμε σύντομα Bye bye. Friends, small talk must take place out. Παρακαλώ, οι κουβέντες παρακαλώ εκτός της αίθουσας. Να επαναλάβω. Κύριε Κάσα, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάσα μου, σας ευχαριστώ για την προσπάθεια την οποία κάνατε με την τελευταία έκθεση. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική για μας νομίζω παρουσίαση και θα δώσω το λόγο στον κύριο Λένερτς. Δημιουργία μιας εποπτικής αρχής εργασίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το επόμενο θέμα λοιπόν η ελευθερία του να κυκλοφορούν, εν πάση περιπτώσει, οι Ευρωπαίοι πολίτες να εργάζονται ή να σπουδάζουν σε άλλες χώρες είναι το βασικό πλεονέκτημα και επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και σε σχέση με την καταπολέμηση του αποκλεισμού, την ελεύθερη κυκλοφορία και τη δίκαιη κυκλοφορία να προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, να προλαμβάνεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού και επίσης να αντιμετωπίζονται γενικότερα τα θέματα της ελεύθερης διακίνησης. Εγώ έρχομαι από την ωραιότερη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα στα σύνορα ε, της ε, Γερμανίας και της Ολλανδίας και πράγματι θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της Ένωσης να επισκέπτονται τις περιοχές αυτές. Απαιτείται λοιπόν να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία της ελεύθερης διακίνησης. Πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες, σαφείς κανόνες, αυστηροί κανόνες. Έχουν γίνει αρκετά. Ε, υπάρχει η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, υπάρχουν σε εκκρεμότητα και άλλοι κανόνες, ε, αλλά οι κανόνες αυτοί στερούνται παντελώς σημασίας αν δεν εφαρμόζονται με ορθό τρόπο. Ε, έτσι μόνο θα πετύχουμε την ελεύθερη διακίνηση. Όσο οι πολίτες γίνονται όλο και πιο κινητικοί, πάνω από 17 εκατομμύρια εργάζονται και κατοικούν σε διαφορετικά κράτη-μέλη, απαιτείται η σωστή εφαρμογή των κανόνων και εδώ η Ευρωπαϊκή Αρχή έχει νόημα. Η πρότασή μου αυτή ε, υποστηρίζει λοιπόν την δημιουργία μιας τέτοιας ε, υπηρεσίας. Γιατί μας λείπει. Η αρχή αυτή θα πρέπει να έχει ε, σαν επιχειρησιακή εντολή την σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας. Καταρχάς ε, εφαρμογή των κανόνων και νομίζω ότι το να υπάρχει και θέμα ε, αποστολής που να αναφέρεται στην ενημέρωση ας πούμε ή στην ε, έβρεση θέσεων απασχόλησης είναι κάτι το περιττό στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να είναι οι μεμονωμένοι πολίτες ενήμεροι φυσικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Αλλά νομίζω ότι για λόγους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας η παροχή αξιόπιστων επικυροποιημένων και προσβάσιμων πληροφοριών δεν θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα της αρχής αλλά να γίνεται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με την δημιουργία των μονοαπευθυντικών θηρίδων, ενώ η αρχή θα πρέπει να ασχολείται με τον βασικό της στόχο, δηλαδή την εφαρμογή των ρυθμίσεων δικαίου. Απαιτείται επίσης να έχουμε και τις αρμοδιότητες και τα μέσα που είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Δεν χρειαζόμαστε εμείς εδώ ε, κάτι το ε, τεχνητό και αδύναμο. Δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε στον εθελεντικό χαρακτήρα. Ε, νομίζω ότι αυτό μόνο συμπληρωματικά μπορεί να υπάρχει. Νομίζω ότι μόνο όταν συνεργαστούμε όλοι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Και νομίζω ότι ο διαιτητικός ρόλος της αρχής μπορεί να περιλαμβάνει ίσως και την ε, ακριβώς την διαιτησία και την έβρεση λύσης σε εργασιακά θέματα. Να υπογραμμίσω λοιπόν ότι εγώ προσπάθησα να κρατήσω μια κάποια ισορροπία ανάμεσα στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και την αρχή της επικουρικότητας από τη μία και την επιθυμία δημιουργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιας υπηρεσίας λειτουργικής. Ελπίζω να κατάφερα να ισορροπήσω τα δύο. Ελπίζω καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας την ισορροπία αυτή να την διασώσουμε. Η επίτροπο Τάισεν ε, θέλει να ξεκινήσει η συνεργασία αυτή ήδη από το 2019. Θέλω και εγώ να συμμεριστώ τη φιλοδοξία αυτή. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Έχουμε ήδη κάνει αρκετές συνεδριάσεις με εκπροσώπους της Επιτροπής, με εμπειρογνώμονες από πανεπιστήμια Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε την συνεργασία αυτή και να μπορέσει να καταστεί λειτουργική το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή των σοσιαλιστών. Πυρίνσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. πράγματι χρειαζόμαστε μια τέτοια Ευρωπαϊκή Αρχή για δύο λόγους. Καταρχάς, ο υπάρχον συντονισμός ανάμεσα στις εθνικές αρχές θα πρέπει να βελτιωθεί και η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών πρέπει να βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρξει μια δίκαιη κινητικότητα και σωστή λειτουργία της αγοράς της εσωτερικής και της αγοράς εργασίας σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες βλέπουμε εμείς κάποιες βαθιά άδικες ε, πρακτικές ε, όπως ε, φιλετικές διακρίσεις, εκμετάλλευση, στρέβλωση των κανόνων που παραβιάζουν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και απαιτούν άμεση δράση. Δεύτερον, διεχόμαστε με ικανοποίηση την πρόταση του μηνός Μαρτίου από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δημιουργία μια τέτοια υπηρεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέπει τη σωστή συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες εθνικές αρχές <coughs> και η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου να γίνεται με σωστό τρόπο. Πρέπει να ενισχύσουμε τις αρχές λοιπόν της υπηρεσίας αυτής και να μπορεί να στηρίζει τις αποκοινού δραστηριότητες των εθνικών αρχών όπως επίσης και τους κανόνες λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρήζει περαιτέρω βελτίωσης και θα πρέπει να στοχεύσει κάπως καλύτερα τις αρμοδιότητες και τις προοπτικές της να επιλεγούν από τις κατάλληλες δομές ή κατάλληλες ενέργειες και δράσεις. Τέταρτον, η πρόταση την οποία μας κάνει ο κύριος Λένερτς, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για τη δουλειά την οποία έκανε, είναι μια καλή βάση για την εκκίνηση των εργασιών μας. υποστηρίζει όπως είπαμε την δημιουργία μιας τέτοιας αρχής και θέλει με συγκεκριμένες αλλαγές να την καταστήσει λειτουργική έτσι ώστε να βελτιωθεί η κινητικότητα. Υπάρχουν δύο θέματα όμως τα οποία δημιουργούν αμφιβολίες και τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Καταρχάς η εμβέλεια δεν θα πρέπει να περιορίζεται ε, μόνο στους αποσπόμενους εργαζομένους. Και δεύτερον, η, επίμονη συγγνώμη, στην ε, επιβολή και τον σεβασμό των κανόνων ίσως να μην ε, θέτει το βάρος εκεί που πρέπει, δηλαδή στη συνεργασία των εθνικών υπηρεσιών. Πρέπει να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Νομίζω ότι αν εμείνουμε προς τη μία κατεύθυνση μόνο, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Ε, κάποιες πιθανές τέτοιες αλλαγές μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στη διαδικασία έγκρισης. Εμείς θέτουμε σαν προτεραιότητα για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής, την διευκρίνηση και τον καθορισμό του συνόλου των στόχων και του πεδίου των στόχων που θα έχει ε, γιατί εδώ υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τις ίδιες νομικές δεσμεύσεις τις οποίες αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν μιλάμε για τους πολίτες, μετακινούμενους πολίτες, οι συνοριακούς πολίτες, μεθοριακούς εργαζόμενους, γενικά υπάρχει μια μικρή σύγχυση εδώ. Μιλάμε για την κινητικότητα συνολικά της αγοράς εργασίας. Υπάρχουν επίσης διαφορές νομικά κείμενα σχετικά με τους ορισμούς των ιδίων δάσεων και ενεργειών και θα πρέπει όλα αυτά να διευκρινιστούν στον κανονισμό, όπως επίσης και οι νομοθετικές πράξεις που θα τον διέπουν. Ο στόχος όμως ε, της συγκεκριμένης ε, δραστηριότητας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Οι προτεραιότητες μας λοιπόν είναι να δώσουμε στην αρμόδια αρχή τις αρμοδιότητες που θα βοηθήσουν την πλήρη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και της κινητικότητας των εργαζομένων. Και δεύτερον να πετύχει μία ισορροπία ανάμεσα στις εθνικές αρχές για τη σωστή εφαρμογή των κανόνων. Η αρχή αυτή θα πρέπει να ενισχύσει και να συνδράμει τις εθνικές αρχές και θα πρέπει να έχει και τον δικό της ξεκάθαρο ρόλο στην αξιολόγηση των κινδύνων και επίσης σε τομείς όπως η διαιτησία. Θα πρέπει να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες κοινοτικές δομές ε, και να είναι σε θέση να κάνει έρευνες και μελέτες στον τομέα της κινητικότητας των εργαζομένων. Πρέπει επίσης να έχει μια οργανωτική δομή. Δε, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες εδώ, θα πρέπει να τονίσουμε τρεις πλευρές. Πρώτον, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε επίπεδο ηγετικό θα πρέπει να έχει μια τέτοια δομή που να επιτρέπει την άμεση συνεργασία με τις εθνικές αρχές και την άμεση ε, ανείχνευση, αν θέλετε, των παραβιάσεων των κοινοτικών κανόνων. Εάν λοιπόν συμβεί κάτι τέτοιο, θα επιτραπεί να λειτουργήσει σωστά η υπηρεσία αυτή και χωρά, ε, χωρίς περιτά προβλήματα και επιβαρύνσεις. Υπάρχει ένα δίκτυο, αν θέλετε, επιτροπών, μονάδων και υπηρεσιών που ασχολούνται με το θέμα της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου στον τομέα της κινητικότητας. Δημιουργούνται λοιπόν παρανοήσεις, είναι δύσκολο να ξεκαθαρίσουμε και να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, κάτι το οποίο θα ήταν όμως απαραίτητο. Και τρίτον, η πλατφόρμα η οποία προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να γίνει δεκτή γιατί δεν περιλαμβάνει ε, πλήρως τις αρμοδιότητες τις οποίες θα έχει η υπηρεσία αυτή. η πλατφόρμα θα πρέπει να μην ελέγχεται απόλυτα από την αρμόδια αρχή, αλλά να είναι ένας χώρος επικοινωνίας ε, που θα επιτρέπει την βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Θα πρέπει να δούμε μια τριμερή δομή, όπως ακριβώς γίνεται σε αντίστοιχους άλλους οργανισμούς στον ίδιο χώρο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι αυτό το οποίο λειτουργεί χωρίς σοβαρά προβλήματα σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να λειτουργήσει και χωρίς πρόβλημα και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Σχετικά τώρα με την ομάδα των εμπλεκομένων συμφερόντων, θα πρέπει να καλύψουμε φυσικά και τους ε, κοινωνικούς εταίρους, για να αποφεύγεται μέσω των μετακινήσεων η εκμετάλλευση η κοινωνική των εργαζομένων. Ταυτόχρονα απαιτείται περαιτέρω προετοιμασία. Δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Μέχρι το 2019 ο χρόνος είναι μια προθεσμία την οποία δεν μπορέσαμε να παρατείνουμε και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο δραστήριοι μπορούμε για να καλύψουμε το μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας. Να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες και ποιες είναι οι προσδοκίες των πολιτών. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Νομίζω ότι άξιζε να επιμείνω σε λεπτομέρειες λόγω της φύσης της συγκεκριμένης προσπάθειας. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κύριε Τρεμπέσιος τώρα από τους ε, ε, μεταρρυθμιστές συντηρητικούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Η έκθεση για την αναφορά της ε, Κομισιόν για τις ε, αρχές των πολιτικών εργασίας ε, υποστηρίζει τις ενσυχίες του ELA για, για τους πολλούς φορείς και τις υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν σε μια γενική υπηρεσία ομπρέλα έτσι ώστε να επιτύχουμε μια επιτάχυνση της διαδικασίας. Αυτό καταρχάς ακούγεται καλό. Στο δεύτερο βήμα ωστόσο οι υπάρχουσες αρχές και τα διάφορα βήματα θα πρέπει να διαλυθούν κατά κάποιο τρόπο γιατί αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν διπλές δομές στην Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Ας πούμε, έχουμε την δημιουργία νέου πόρταλ πληροφορικής, το οποίο μπορεί να βρίσκεται σε ανταγωνισμό με τις υπάρχουσες δομές. Και δεν είναι απόλυτα σαφές επίσης αυτό το νέο πόρταλ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς ακριβώς θα είναι προσβάσιμο και ποια προσθέμενη αξία θα έχει. Επίσης, από πολλές εθνικές κυβερνήσεις υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο εδώ ισχύει και μπορεί να παραμείνει ισχύει η αρχή της επικουρικότητα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι νέε δομέ εντός του υπάρχοντος ε, προπολογισμού θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν. Εάν ε, θέλουμε τώρα να έχουμε μια προσθέμενη αξία ευρωπαϊκή, θα πρέπει να δούμε το γενικό συνολικό κόστος. Οι νέε δομέ κατά δική μας την άποψη, θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικέ και να λειτουργούν καλύτερα από ό,τι παλιές. Επίση, δεν θα πρέπει να υπάρξει ε, ε, ανακατανομή των αρμοδιοτήτων, σίγουρα όχι μέσω τη ε, διαμεσολάβηση. Αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτική όταν μιλούμε για την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατών μελών. Για τις τρίτες χώρες επίσης και τους ποιητικούς τριτοχωρών θα υποβάλω εγώ κάποιες ε, ε, τροπολογίες για την ε, άδεια παραμονής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες από, τις, από τους κανόνες που ισχύουν για, τους, για την παραμονή των Ευρωπαίων πολιτών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και επίσης μια παρατήρηση για την προσθήκη των δεδομένων. Ξέρουμε ότι οι δημόσιες αρχές ε, είναι αρκετά ευαίσθητε ό,τι αφορά τι ευάλωτε σχετικά με τι ε, επιθέσει στο διαδίκτυο και ο ELA έχει μια δυνατότητα αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξουν κάποιε προβλέψει για την προστασία αυτών των δεδομένων. Και τέλο, να μιλήσω για την αυτόματη παράταση αυτή της πενταετία ε, αποθήκευση των δεδομένων. Τα επόμενα χρόνια οι ε, ευρωπαϊκές αρχές θα ασχοληθούν με την οδηγία για τις αποσπάσεις και βεβαίως ε, θα αλλάξουν τα πράγματα και με υπό το φω του Brexit. Αυτές οι νέε δομέ θα πρέπει να ανταποκριθούν στι νέες προκλήσει που είναι σημαντικέ και πρέπει αυτό να το εξετάσουμε. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα αξιολογήσουμε εντό ενό συγκεκριμένου χρονικού διαστήματο. Χαίρομαι για τη συνεργασία με τον εισηγητή και θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο επικοδομητική γίνεται. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Η Μάριαν Χάρκιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όλοι στην Επιτροπή μα και στο Κοινοβούλιο γενικώ ε, είναι υπέρ των προτάσεων που θα οδηγήσουν σε καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και αν δούμε τον κατάλογο προκλήσεων που μας παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή έχουμε ανεπαρκή υποστήριξη ή καθοδήγηση των ατόμων, δυσκολίες στις διασυνοριακές περιπτώσεις ή ανεπαρκής ικανότητα σε εθνικό επίπεδο για την οργάνωση συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών ε, σε διασυνοριακό επίπεδο. Και είναι ενδιαφέρον ότι περάσαμε από τον όρο κινητικότητα στον όρο δίκαιη κινητικότητα τα τελευταία χρόνια. Γιατί λέμε ότι η ελεύθερη διακίνηση προσώπων είναι θεμελιώδης αρχή, αλλά χαίρομαι που βάζουμε και το επίθετο δίκαιο στην κινητικότητα. Και για να εξασφαλίσουμε αυτή την ελεύθερη διακίνηση, ε, χρειαζόμαστε κάποιους κανόνες για να διαφυλάξουμε και την δίκαιη κινητικότητα. Αυτό προϋποθέτει ενημέρωση, ε, υποστήριξη, παροχή συμβουλών, συνεργασία μεταξύ των οικειών και συμφωνώ με τον εισηγητή κάτι τέτοιο προϋποθέτει και κάποιους μηχανισμούς για την εφαρμογή, επιβολή αυτών των κανόνων. Οπότε η ερώτηση που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι κατάλληλος μηχανισμός, κατάλληλος φορέας ε, και θα ανταπεξέλθει στην αποστολή του. Δηλαδή θα υλοποιήσει όλους αυτούς τους στόχους, θα έχει τις εξουσίες να το καταφέρει, θα έχει τους σπόρους, την, τις ικανότητες. Αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στην Επιτροπή και όπως ε, ε ρώτησαν και άλλοι προλαλήσαντες, προσφέρει μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ξέρω ότι παρέχουν αρρωγή κάποια κράτη-μέλη και κυρίως οργανώσεις σε κράτη-μέλη ε, και υποστηρίζουν την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά προσεκτικά. Πάντως θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λενάρς, τον εισηγητή μας για το έργο του. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη θέση του. Είπε ότι ε, η βασική αποστολή της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας είναι η επιβολή των κανόνων και είπε μάλιστα ότι δεν θα πρέπει η ανάμειξη των κρατών μελών, η εμπλοκή να είναι οικειοθελής, προαιρετική, παρά μόνο υπό εξαιρετικές συνθήκες. Θα εξετάσουμε τις προτάσεις του, είναι ε, αρκετά σημαντικά αυτά τα θέματα και ίσως ε, αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες. Πάντως, η δική μου θέση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα πρέπει να ε, προσφέρει ουσιαστική προστιθέμενη αξία και θα πρέπει να έχει την εξουσία, την αρμοδιότητα, την ικανότητα, δεν ξέρω τι ορολογία θα χρησιμοποιήσουμε για να το κάνει. Επίσης, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην εκτοπίσει ούτε να υποκαταστήσει η ΕΛΑ ε, το αξιόλογο έργο άλλων φορέων, όπως τη πλατφόρμα κατά της εργασία. και φυσικά ο εξορθολογισμό είναι πολύ σημαντικό στόχο, αλλά προσοχή να μην πάει χαμένο το μέχρι τώρα έργο που έχουν κάνει άλλοι φορεί. Ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή και ε, αδειμονώ να λάβω μέρος στις ε, πολλαπλές συνεδριάσεις που έχει προγραμματίσει με τους και οδησηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή για την παρουσίασή του. Να είμαι ειλικρινής, εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο να υπάρξει μια σαφή θέση. Ε, είναι δύσκολο να δούμε ποια είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία. Από την άλλη έχουμε μια ολόκληρη σειρά προκλήσεων μπροστά μας. Αν δούμε ποιο είναι το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα της ελεύθερης διακίνησης του εργατικού δυναμικού, το θέμα είναι ότι η εσωτερική αγορά χρησιμοποιείται από τους εργοδότες για να πιέζουν ε, τους εργαζομένους σε τοπικό επίπεδο. Συνεπώς ε, έχει σημασία να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορεί να κάνει η νέα αυτή αρχή. Αν δούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην αύξηση της κινητικότητας. Θέλει να καταστήσει την κινητικότητα ευκολότερη. Η ομάδα μας όμως πιστεύει ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε άλλο θέμα. Ε, να δώσουμε έμφαση στη δίκαιη κινητικότητα για να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό dumping. Και επίση να εφοδιάσουμε τι εθνικέ αρχέ με συντονιστική ικανότητα ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν σε περίπτωση που γίνεται κατάχρηση τη εσωτερική αγορά για να ασκηθεί πίεση στι εργασιακέ συνθήκε. Οπότε οι τροπολογίες μας έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Καταρχήν θα πρέπει να βελτιώσουμε όχι την κινητικότητα, αλλά την αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ για να έχουμε μεγαλύτερη μισθολογική ισοτιμία. Επίσης να δώσουμε το λόγο στους κοινωνικούς εταίρους δεν θα πρέπει να τους περιορίζουμε μόνο σε συμβουλευτικό ρόλο. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργοί, όπως το κάνουν σε πολλά και θα πρέπει να έχουν αποφασιστικό ρόλο στο έργο της νέας αρχής, της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Επίσης, θα πρέπει να τους δώσουμε το σωστό ρόλο και τη θέση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας, γιατί και εκεί υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Σε μερικές χώρες συμμετέχουν τα συνδικάτα, σε άλλες ε, ε, εφαρμόζεται άλλο σύστημα. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία δεν θα πρέπει να καταστρέψει, να υπονομεύσει ότι ήδη λειτουργεί εύρυθμα σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να στηρίζει τι κατάλληλε εθνικέ ρυθμίσει και να βελτιώνει τα πράγματα. Επίση, δεν θα πρέπει να απορροφά ε, πόρου που προορίζονται για τα κράτη-μέλη. Τι θα γίνει με το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν αποσπάσουμε ε, κάποιους από το Συμβούλιο επιθεώρηση για να του βάλουμε σε υπολογιστέ, να δουλεύουν μπροστά σε υπολογιστέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι αυτή η σωστή αξιοποίηση των πόρων. Όπω καταλάβατε, είμαστε αρκετά επικριτικοί απέναντι στην πρόταση, αλλά είμαστε πρόθυμοι για διάλογο επικοδομητικό προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια πραγματική προστιθέμενη αξία και να ενισχύσουμε και το ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει εκπρόσωπος των Πρασίνων. Όχι, οπότε πάμε στην EFTD. Έχουμε εκπρόσωπο της ομάδας EFTD. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Από το ENF. Ούτε από το ENF. Ευχαριστώ τότε. Η κυρία Σόιντροβα ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όσους έχουν κάποιες αμφιβολίες για αυτή τη νέα αρχή εργασίας. Δεν θα είναι ακριβώς υπηρεσία, θα είναι αρχή ε, και θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν τι θέλουμε ακριβώς. Θέλουμε μια νέα αρχή με ισχυρές αρμοδιότητες και εξουσίες ή θέλουμε μια υπηρεσία η οποία θα έχει μάλλον συντονιστικό ρόλο. Εγώ καταλαβαίνω ότι χρειαζόμαστε μια αρχή ή τέλο πάντων ένα είδο υπηρεσίας που θα βοηθάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την, για την εφαρμογή του δικαίου εργασίας και για την διεξαγωγή των ελέγχων της εφαρμογής αυτού του δικαίου. Και βεβαίω ε, που θα επιβάλλει και ένα γενικό πλαίσιο. Αυτό είναι ο πυρήνα τη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται δηλαδή να απασχολήσουμε και νέου υπαλλήλου κτλ. Τη δουλειά τη. Ε, η δουλειά αυτή τη υπηρεσία θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε και αυστηροί σε ό,τι αφορά την αρχή τη επικουρικότητα. Θεωρώ επίση ότι η αρχή αυτή όπως είπαμε στη νέα διοργανική συμφωνία, η έδρα αυτή της, ε, αυτής της αρχής θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα νέο κράτος μέλος. Και επίσης ε, να πω ότι μιλούμε για μία υπηρεσία, αλλά δεν θα είναι υπηρεσία αυτή ε, όπως την ξέρουμε. Ας είμαστε προσεκτικοί, γιατί οι υπάλληλοι θα πληρώνονται. Δεν ξέρω η Κομισιόν πώς σχεδιάζει να το διαχειριστεί όλο αυτό. Εγώ προσωπικά περιμένω αν ε, αστραφεί μια υπηρεσία, μια επιχείρηση ας πούμε σε αυτή την ε, ε, υπηρεσία και θέλει να ξέρει ποιες είναι ας πούμε οι υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσει, θα πάρει δωρεάν τις πληροφορίες από αυτή την αρχή, τις πληροφορίες που χρειάζεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε κάνω έκκληση να είμαστε προσεκτικοί με, την, ε, με τις αρμοδιότητες που έχουν τα κράτη-μέλη. Να τις ενισχύσουμε. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει δικαίωμα να μπορεί να εκπροσωπεί, ε, να εκπροσωπείται σε αυτή την ε, υπηρεσία, σε αυτή την αρχή. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε το λόγο του κ. Διντιέ. Ε, βλέπουμε ότι ε, υπάρχει μια δυσπιστία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πολλούς Ευρωπαίους πολίτες και ιδιαίτερα είναι καχύποπτη επένδυση στη δημιουργία νέων φορέων ή αρχών ή οργανισμών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αντίδραση της κοινή γνώμης, γιατί θα προβληματιστεί η κοινή γνώμη κατά πόσο είναι χρήσιμη ή απαραίτητη μια τέτοια νέα δομή, μήπως θα υποκαταστήσει τα κράτη-μέλη, ποιες θα είναι οι εξουσίες, οι αρμοδιότητές της, μήπως έχει υπερβολικές αρμοδιότητες. Είναι εύλογες όλες αυτές οι ανησυχίες και θα πρέπει να διαλύσουμε κάθε ασάφεια. Πάντως πιστεύω ότι η κοινωνική Ευρώπη χρειάζεται μια ουσιαστική ευρωπαϊκή αρχή εργασίας για να καταπολεμήσει τις κοινωνικές απάτες, τον αθέμητο ανταγωνισμό και όλες τις αδικίες που μερικές φορές ε, δημιουργούνται από την κινητικότητα. Και αυτή η αρχή θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχει ως αποστολή την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων εργαζομένων για να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Και θα πρέπει να έχει και τους πόρους για να το κάνει. Γιατί είναι ε, νομοποιημένη και θεμητή η αρχή εργασίας και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι παρόν ε, στέλνοντας εμπειρογνώμονες στο Διοικητικό Συμβούλιο, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Αλλά θα πρέπει και ο προϋπολογισμός να είναι φιλόδοξος, φυσικά όχι εις βάρος άλλων κοινωνικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπό τον όρο επίσης ότι η αρχή αυτή δεν θα μετατραπεί ε, σε μόνο ε, λόγια. Θα πρέπει να δώσουμε ένα λειτουργικό επιχειρησιακό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Αρχή αλλά το πλαίσιο τη να είναι περιορισμένο, δηλαδή να σέβεται απόλυτα ε, τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Και επίσης θα ήθελα να αποδείξω φόρο τιμής στον συνάδελφο Λάνερς, που με τα σχόλιά του, τη σκέψη του και την πρότασή του, ε, κατάφερε να βρει μια σωστή ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των κρατών μελών και, της, και του καθήκοντος Ευρωπαϊκής Ένωσης για περισσότερη προστασία. Ευχαριστώ κύριο Καλβέ Σόμπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα είμαι λακωνικός γιατί η κυρία Χάρκιν ε, μας παρουσίασε τη θέση των φιλελευθέρων. Ε, συμφωνώ απόλυτα μαζί της και συνεχίζοντας τον ερμό του προλαλήσαντος με τον οποίο συμφωνώ 80% θα ήθελα να πω τα εξής. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Αρχή Εργασία παρεμβαίνει στην κυριαρχία των κρατών μελών. Δεν θα πρέπει έτσι να θέσουμε τους όρους της ε, συζήτησης. Και τότε τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή τι συμβαίνει με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο. Όχι, δεν μιλάμε εδώ για τα κράτη-μέλη. Εδώ με την πρόταση αυτή αναγνωρίζουμε ότι οι αγορές εργασίας των κρατών μελών για πολιτιστικούς, ε, ε, κλιματικούς, γεωλογικούς ή λόγους παράδοσης ή κοινωνικού ιστού, οι, διαφορές, οι αγορές αυτές των κρατών μελών είναι ε, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και δεν υπάρχει τρόπος να αποκαταστήσουμε μια ομοιομορφία μεταξύ των αγορών αυτών που εδώ και αιώνε ολόκληρου λειτουργούν με το δικό του τρόπο. Αλλά έχουμε ταυτόχρονα μια εσωτερική αγορά με πλήρη κινητικότητα. Τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρχει πλήρη κινητικότητα. Και μια σειρά ε, θεμελιωδών ε, προγραμμάτων, ε, προβλημάτων που αφορούν τα ελάχιστα δικαιώματα, του περίφημου κοινωνικού πυλώνα. Και το, το θέμα αυτό ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να ορίσουμε το πλαίσιο και όχι τις λεπτομέρειες της ε, εθνική αγορά εργασία, που γίνεται σεβαστή. Αλλά θέλουμε στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής προοπτικής να λαμβάνουμε υπόψη τη οικονομία κλίμακος, να δίνουμε προσανατολισμό, να ελέγχουμε τη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο που επίση έχει τη θέση του στην ένωμη τάξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης είναι σημαντικό να έχουμε μια τέτοια αρχή. Δεν θα είναι τέλεια, δεν είμαστε θέοι για να κάνουμε τέλεια πράγματα, αλλά προς θα δημιουργήσουμε ένα χρήσιμο όργανο για τον κόσμο, για τους πολίτες, για τους Ευρωπαϊ... Ευρωπαίους εργαζομένους και θα την τελειοποιήσουμε στην πορεία αυτή την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Και η συνέχιση της θα δικαιολογηθεί από τα θετικά αποτελέσματα που θα έχει υπέρ της προάσπισης των ε, θεμελιωδών κοινών δικαιωμάτων. Προσοχή όμως να δώσουμε τις λειτουργίες που περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, του ελέγχου, της ε, δημιουργίας γνωμόνων, της αφομοίωσης των αποτελεσμάτων και να μην τις αναθέσουμε ε, αρμοδιότητες που ήδη έχουν άλλοι φορείς οργανισμοί. Δεν θα ήθελα να καταρτίζει ε, μελέτες η Ευρωπαϊκή Αρχή Η Eurofound, το CEDEFOP, η όσα κάνουν μελέτες. Θέλουμε μια συντονιστική λειτουργία, σίγουρα αυτό χρειάζεται, αλλά όταν μιλάμε για τα προβλήματα των πόρων, σίγουρα θα πρέπει να αποφύγουμε επικάλυψη αποστολών και να δούμε πού ε, χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Αρχή Και χρειάζεται σε πολλά με μονομένα καθήκοντα, αλλά αποφεύγοντας την επικάλυψη με άλλους φορείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλο κανένα θέλει το λόγο. Άλλος κανείς παρακαλώ. Όχι. Οπότε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν υπάρχει κάποιο ε, εκπρόσωπο Γενική Διεύθυνση Απασχόληση που θέλει το λόγο, πολύ ευχαρίστω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ονομάζομαι Ζαν Τόμα από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και θα ήθελα εν συντομία να ε, πω τρία πράγματα. Καταρχήν ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας επιτρέπετε σήμερα να είμαστε εδώ και να λαμβάνουμε μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Ε, είναι όντως πιεσμένο το χρονοδιάγραμμα και όπως είπε ο εισηγητής, ήδη από την αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπέβαλε ένα πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα και εσείς το τηρείτε και χαίρομαι γι' αυτό. Γνωρίζω ότι είναι πολύ ε, στενές οι προθεσμίες, κάτι που μας αναγκάζει σε πολύ έντονη ανασχόληση με το θέμα αυτό και σας ευχαριστώ και για την θερμή υποστήριξη που δείξατε για την πρότασή μας στην έκθεση σας. Φυσικά έχουμε κάποιες διαφορές μεταξύ μας. Θα τις συζητήσουμε από τη στιγμή που θα οριστικοποιηθεί και θα αποσαφινιστεί η εντολή. Και γι' αυτό πραγματικά περιμένουμε με ανυπομονησία τη σχετική συζήτηση. Διαβάσαμε την έκθεση, ακούσαμε τα σχόλια, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διαφορές ε, και φυσικά θα χρειαστούν κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες ε, για τις προτάσεις μας. Καταρχήν, ποια είναι τα καθήκοντα που προβλέπουμε για την Ευρωπαϊκή Αρχή εργασία. Το πρώτο είναι η ενημέρωση. Το έβδομο ε, καθήκον, η έβδομη αποστολή είναι διευκόλυνση, διαμεσολάβηση σε περίπτωση διαταραχών τη αγορά εργασία. Και εδώ έχετε διαφορετική προσέγγιση. Πάντω, ακούσαμε τα σχόλιά σα για τον τίτλο, την προστιθέμενη αξία, να μην γίνει ένας ανίσχυρος ε, φορέας, ξεδοντιασμένος ε, ε, τίγρης, επίσης να μην είναι μόνο φούμαρα, να έχει μια ουσία και να σας πω ότι η πρόταση αυτή είναι ένα πακέτο που εξασφαλίζει και πρόληψη και σωστή εφαρμογή των υφισταμένων κανόνων. Και η Ευρωπαϊκή Αρχή θα προσφέρει Πληροφορίε ενημέρωση και θα βοηθάει και τα κράτη-μέλη να ενημερώνουν σωστά του ενδιαφερομένους. Αυτό είναι τμήμα της πρόληψης των αδικιών. Ευχαριστώ και πάλι θερμά και σας ε, διαβεβαιώ ότι είμαστε πρόθυμοι για συνέχιση της συζήτηση με τον εισηγητή και τους και εισηγητές εννοείται και θα κρατούμε επαφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν είναι το εξή. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών η 17η Ιουλίου. Την επόμενη εβδομάδα, 17 Ιουλίου. 12 το μεσημέρι. Εξέταση των τροπολογιών στις 29 και 30 Αυγούστου. Ψηφοφορία τον Οκτώβριο, 18 Οκτωβρίου. και δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία για την Ολομέλεια. Ο κύριος Λέναρτς, αν θέλετε να προτείνετε την ε, προθεσμία να αλλάξει και να την κάνετε μέχρι αύριο, τόσο το καλύτερο για μένα. πραγματικά θα το ήθελα, λέει η πρόεδρος, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω. Θα μας ανακούφιζε για το καλοκαίρι. Καλώς σας, ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Προστασία των πολιτών οι οποίοι φέρνουν στην ε, επιφάνεια παραβιάσεις του ε, κοινοτικού δικαίου. Ο κύριος Ηλικιώτης είναι εισηγητής, αλλά αντικαθίσταται. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Σιλικιώτη, δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα και μου ζήτησε να σας παρουσιάσω κάποιες από τις παρατηρήσεις του. Το σύνολο της πολιτικής του ομάδας παρακολουθεί τα θέματα αυτά πάρα πολύ κοντά γιατί έχει μεγάλη σημασία ε, να ε, γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται με τους ε, καταγγέλλοντες για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ταυτόχρονα προσπαθήσαμε, λέει ο κύριος Σιλικιώτης, να ενσωματώσουμε όσο λιγότερες τροπολογίες μπορούμε ε, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ακριβώ τις αρχικές μα θέσεις. Καταρχάς υπάρχει η ανάγκη εγγύηση της ανωνυμία. Θα πρέπει να είμαστε ανώνυμοι όταν καταγγέλουμε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Θα πρέπει επίσης ε, να μπορούν να λειτουργούν οι υπάλληλοι οι οποίοι θα προστατεύονται στα πλαίσια της οδηγίας αυτής όταν καταγγέλουν κάτι. Θέλουμε επίσης ένα σημαντικό επίπεδο προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο εισηγητής είναι υπέρ μια κάποιας μορφής οργάνωσης που θα προστατεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο σε όλη την Ευρώπη. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια οριζόντια διαδικασία σε σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Θα μπορούν δηλαδή οι καταγγέλλοντες και εσωτερικά να κάνουν την καταγγελία αλλά και σε επίπεδο δημοσίας αρχής. Ε, τώρα για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να διευρυνθεί έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι πλευρές του δημοσίου συμφέροντος όπως η εργασιακή νομοθεσία που μας ενδιαφέρει εδώ εμάς και επίσης και κάποιες άλλες μορφές στρατηγικής οι οποίες καλύπτουν το δημόσιο συμφέρον. Και τέλος ο ίδιος ο ρόλος των καταγγελόντων αυτών δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι άμεσα εργαζόμενο σε μια επιχείρηση. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος για διαφορετικούς λόγους έχει συμφέρον για το θέμα αυτό. Συνεπώς λοιπόν και σε σχέση με τις προσθήκες θα καταθέσουμε ορισμένες τροπολογίες επιπλέον γιατί θα πρέπει να αποφύγουμε ε, διαδικασίες ιδιαίτερα περίπλοκες. Πάντως πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία μπορούν να καλύψουμε από κοινού. Περιμένω τις προτάσεις σας και ελπίζω στο τέλος να έχουμε μια εξαιρετική γνωμοδότηση για το σύνολο της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων Αρμόδιας επί της ουσίας. Σας ευχαριστώ. Ένας από τους κοιόδης είναι ο κ. Χάσε, τον αντικαθιστά κάποιος, όχι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι Ανεξάρτητα αν τα Panama Papers και τα LuxLeaks ε, καθιστούν αναγκαία την οδηγία αυτή, ξεκαθαρίστηκαν τα πράγματα από τα όσα είπε ο συνάδελφος ε, για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Μιλούμε για εσωτερικό και εξωτερικό σύστημα Σαφέ είναι ότι οι κοινωνικοί εταιρείε στην δημιουργία αυτού του συστήματο θα πρέπει να ε, συμμετέχουν στην όλη διαδικασία σχεδιασμού του. Εδώ νομίζω ότι η έκθεση δεν είναι απόλυτα σαφή για το πώ θα γίνει αυτό. Η πρόταση οδηγία περιλαμβάνει μόνο ένα ε, ε, δίκαιο προστασία για αυτές τις ε, παραβιάσεις στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι θα γίνει. Τώρα, με τις παραβιάσεις κατά των δικαιωμάτων των εργαζομένων, επίσης δεν είναι σαφές το τι θα γίνει. Θα πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν. Γιατί αν μείνουν τα πράγματα όσο έχουν είναι πραγματικό, πραγματικά απαράδεκτα. Η νομική βάση επίσης ε, μιλά για την ενίσχυση της ε, εσωτερικής αγοράς. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ περίεργες καταστάσεις ένας εργαζό, εργαζόμενος μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει ε, παραβίαση του ε, δικαίου, του ε, δικαίου για την προστασία των ζώων, αλλά δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει παραβίαση κατά των δικών του δικαιωμάτων, των εργασιακών. Αυτό πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το καλύψουμε. Νομίζω ότι βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο περιθώριο για διατροποποίησεις, για βελτιώσεις, οπότε χαίρομαι πραγματικά για τη συνεργασία που θα έχουμε με τους συναδέλφους. Αυτά από μένα και ευχαριστώ. Thank you. Ε, Mr. Hodge, representing... Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος ε, του ECR. Ε, Ο κύριος ε, ο προλαλής σας αναφέρθηκε στα LuxLeaks και στα έγγραφα του Παναμά. Να προσθέσουμε και το Dieselgate, το σκάνδαλο με την Cambridge Analytica και την υπόθεση Τζάκο κατά της ε, Μολδαβίας. Είναι εμ, αποδείξεις ότι χρειαζόμαστε τους καταγγέλλοντες. Πολλό δε μάλλον όταν έχουμε παγκοσμιοποίηση και όταν έχουμε αυτή την ε, προσήλωση πολλών στο κέρδος και στη, στο χρήμα. Και στο μέτρο που ε, η οικονομία και το κέρδος ε, θα κυριαρχούν στον κόσμο, χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο τους καταγγέλλοντες που καθοδηγούνται μόνο από το δημόσιο αγαθό και το, αγαθό, το καλό της κοινωνίας. Θα πρέπει να βρούμε ένα λοιπόν ευρωπαϊκό τρόπο για να προστατεύσουμε αυτούς τους καταγγέλλοντες. Έχω κάποιες παρατηρήσεις όμως για την οδηγία αυτή και κάποιες επιφυλάξεις. Για το πρώτο άρθρο, για παράδειγμα, εκεί που αναφέρεται η προστασία σε κάποιους τομείς, θα πρότεινα να διευρύνουμε τον αριθμό των τομέων, ώστε να περιλάβουμε και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, να αναφέρουμε και τα, τον κίνδυνο βασανιστήριων Επίσης το άρθρο 4 αναφέρονται κάποιοι, κάποιοι δημόσιοι φορείς και το όριο των 10.000 κατοίκων. Ε, γιατί να εξαιρέσουμε μικρότερες δήμους ή κοινότητες από την οδηγία. Γιατί αν έχουμε δήμους κάτω των 10.000 ε, είναι στο απειρόβλητο τέτοιου είδου μικρότερες κοινότητες. Μπορεί να έχουν φυσικούς σπόρους, μπορεί να έχουν κάποιο φυσικό πλούτο, οπότε να γίνονται και εκεί κάποιες ατασταλίες ή παρατυπίες. Επίσης, στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι οι καταγγέλλοντες υπόκειται στην προστασία ε, σε, ε, από εξωτερικούς παράγοντες μόνο όταν έχουν εξαντλήσει τους εσωτερικούς διάβλους. στις ε, ενέργειες όμως που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και έχουμε ε, δύο επιχειρήσεις που ε, ανταγωνίζονται, οι εσωτερικές δράσεις δεν θα αποφέρουν αποτελέσματα και θα εκθέσουν τον καταγγέλλοντα σε υπερβολικό κίνδυνο. Οπότε και αυτό το θέμα θα πρέπει να το εξετάσουμε. Θα ήθελα και να προσθέσω και ένα δικό μου σχόλιο η Πολωνία θα υποστηρίξει αυτή την πρόταση και αυτό το σχέδιο και θα ήθελα να πω ότι εμείς στην Πολωνία θα έχουμε μεγάλη δυσκολία να έχουμε μια συνολική προστασία των καταγγελόντων, γιατί έχουμε ήδη πολύ καλή εμπειρία με τους ε, πληροφοριοδότες που ήταν ε, καταδότες όμως ε, κατά τη διάρκεια του Σοβιετικού ζυγού και έχουμε δυστυχώς ε, πολύ ε, κακές εμπειρίες με αυτούς τους πληροφοριοδότες, τους καταδότες ε, και σε ένα, προ... ένα σχέδιο προστασίας καταγγελόντων θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια διαπαιδαγώγησης κοινωνίας για να ξεπεράσουμε την παραδοσιακή μας καχυποψία. Γιατί σε, πολλοί, σε άλλες χώρες μπορεί ένας καταγγέλων να, να θεωρείται ως αφανής ήρωας, αλλά στην Πολωνία, λόγω της εμπειρίας που είχαμε από το Σοβιετικό καθεστώς, ένας καταγγέλων για μας είναι πληροφοριοδότης, είναι καταδότης. Ε, είναι δύσκολο λοιπόν να κάνουμε αυτή τη μεταστροφή. Και μάλιστα ε, έχουμε εξετάσει ένα νομοσχέδιο για την προστασία των καταγγελόντων, αλλά σας Ζητώ να λάβετε υπόψη πόσο δύσκολο είναι αυτό το θέμα για του Πολωνού λόγω τη ιστορία μα. Πάντω σα διαβεβαιώ ότι θα υποστηρίξουμε τη σχετική οδηγία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ενδιαφέροντα αυτά που μα είπατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είσαστε η μόνη πρόεδρος που ξέρει ότι το επίθετό μου δεν είναι τουμ, αλλά τόμ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Να κάνω κι εγώ κάποια σχόλια. Πρέπει να πω ότι νιώθω λίγο άβολα γιατί δεν είμαι στην ίδια γραμμή με τους προηγούμενους ομιλητές. Είναι διαφορετικές οι εμπειρίες μας μάλλον και οι διαφορετικές εμπειρίες που έχω εγώ ε, σε σχέση με τα όσα είπε και ο Πολωνός συνάδελφος. Ε, εγώ έζησα το καθεστώς που ενθάρρυνε τις ε, καταδόσεις και μη ε, φανταστείτε ότι αυτό ήταν, ε, γινόταν μόνο για πολιτικούς σκοπούς. Στη Σοβιετική Ένωση υπήρχαν θέματα διαφθοράς όπως και παντού και πραγματικά είμαι πεπισμένη ότι αν ε, ε, ε, υποκινήσουμε αυτή τη διαδικασία θα δημιουργηθούν πολύ περίεργες καταστάσεις γιατί οι άνθρωποι δημιουργούν τις σχέσεις τους με βάση την εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, θεσμικών οργάνων και πολιτών. Όλα αυτά θα πρέπει να βασίζονται στην εμπιστοσύνη. Και είμαι σίγουρη που υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι όντως απαραίτητη η κατάδοση σε εισαγωγικά. Αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό μόνο όταν υπάρχουν πολύ σημαντικά συμφέροντα που διακυβεύονται. Να μην διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή χωρί καλού λόγου τη ε, οδηγία αυτή, οπότε δεν μπορώ να υποστηρίξω την πρόταση να ε, διευρυνθεί η οδηγία αυτή και στην παραβίαση εργασιακού δικαίου. Γιατί εκεί μπορεί να μπουν πολλές πτυχές. Ο πληροφοριοδότης ε, δεν θα πρέπει να είναι ανώνυμος. η ανώνυμη κατάδοση είναι ανήθικη. Ο πληροφοριοδότης θα πρέπει πάντα να δίνει το όνομά του στην αρμόδια αρχή. Μπορώ να δεχτώ την ε, διάταξη για την πρόσταση των δεδομένων, αλλά όχι την ανωνυμία. Η ανώνυμη κατάδοση απαγορευόταν και στη Σοβιετική Ένωση. Δεν το συγκρίνω, δεν συγκρίνω τις δύο ενώσεις, απλώς μιλώ για τις εμπειρίες που έχουμε και που έχω, ε, τον οποίο έχω υπάρξει μάρτυρας η κατάδοση μπορεί να είναι και δικαιολογημένη και όχι. Το να προστατευτεί σε κάθε περίπτωση ο ε, πληροφοριοδότης είναι σωστό. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να καταστρεφεί η φήμη μια εταιρεία ενός οργανισμού εν μία ανοιχτή. Οπότε υποστηρίζω την πρόταση της, ε, τη θέση της Κομισιόν. Προτείνει μια διαδικασία για να μελετήσουμε την ε, έκθεση πρώτα αυτή εσωτερικά μια εταιρεία ή ένας οργανισμό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει επίση την έκθεση και αν μπορεί να λύσει και το πρόβλημα. Και επίσης η εσωτερική ε, διαδικασία ελέγχου για του ε, πληροφοριοδότε μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου ένα εξωτερικό ελεγκτή μπορεί να, είναι, να βασιστεί στι ε, καταγγελίε κάποιων μη ικανοποιημένων εργαζομένων, α πούμε. Επίσης, οι δομές που θα δημιουργηθούν δεν θα πρέπει να ε, δημιουργούν επικαλύψεις με υπάρχοντες ε, ε, οργανισμούς, όπω α πούμε το Ελεκτικό Συνέδριο ή η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου. Και τέλος, αν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε για διεύρυνση των καλών πρακτικών που δεν αναφέρονται μεν και σε χώρες που έχουν ε, συμφωνίες σύνδεσης μαζί μας. Μιλούμε για ευρωπαϊκά χρήματα, για χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου, οπότε καλό θα ήταν να συμπεριλάβουμε και τους συμμάχους, ας πούμε, τους εταίρους μας που παίρνουν πολύ μεγάλα ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας είμαστε λοιπόν όλοι πολύ προσεκτικοί όταν δουλεύουμε σε τέτοια σχέδια οδηγία για να βρούμε την ισορροπία. Να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των, ε, των ε, εμπλεκόμενων φορέων και να προστατεύσουμε και τα συμφέροντα της Ένωσης. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Λάμπερτς. Θέλετε το λόγο, κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Νομίζω ότι έχουμε μια καλή βάση για να ξεκινήσουμε. Με ενδιαφέρουν πολύ οι οπτικές των συναδέλφων σε ό,τι αφορά τις εμπειρίες που έχουν και άρα πώς ε, ε, βλέπουν αυτοί το πολύ σημαντικό αυτό θέμα και πώς θα πρέπει να το εξηγήσουμε, πώς θα πρέπει να το παρουσιάσουμε σε σχέση με τα συμφέροντα που προσπαθούμε να προστατεύσουμε εδώ. Τα παραδείγματα λοιπόν που αναφέρθηκαν ήδη για τα πρόσφατα θέματα, είτε ήταν το LuxLeaks, είτε ήταν τα τα Panama Papers ή τα Cambridge Analytica. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά δημιουργούν τεράστιο ενδιαφέρον και στο ευρύ κοινό και πραγματικά θίγουν πολύ θεμελιώδη ερωτήματα για το πώς λειτουργούν τελικά τα πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι για τη δική μας την ομάδα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νομοθετικό κείμενο και θέλουμε να προχωρήσει και επιτέλου προχωρεί από την πλευρά τη Κομισιόν. Συμμερίζομαι τι ανησυχίε για την νομική βάση και την διεύρυνσή τη σε θέματα εργασιακού δικαίου. Κατανοώ αυτό που ακούστηκε ότι υπάρχουν δύο άφορε αρχέ, αλλά όταν ε, μελετούμε ε, βαθιές και συστημικές καταχρήσεις, παραβιάσεις, ε, γιατί να εξαιρούνται αυτές, αυτοί οι τομείς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κακόβουλη κατάδοση, ε, κάποια κράτη-μέλη ή τα κράτη-μέλη γενικώ θα έπρεπε να έχουν ήδη μέτρα για εναντίον ατόμων που επίτηδε προσπαθούν να καταστρέψουν τη φήμη άλλων συμπολιτών ή, εργαζο... ή ε, ε, επιχειρήσεων. Οπότε δεν βλέπω να υπάρχει λόγος να μπουν έξτρα κυρώσεις όπως προτείνεται εδώ. Το θέμα τώρα της προστασίας ε, εναντίον αντιπίνων θα πρέπει να διευρυνθεί και σε αυτούς που βρίσκονται κοντά στον ε, ε, πληροφοριοδότη, όχι μόνο στο άτομο αυτό καθ' αυτό, και μετά κάποια άλλα που, θέματα που θέλουμε να δείξουμε για την παροχή πληροφοριών και προς το άτομο που κάνει την καταγγελία, ώστε μετά την καταγγελία, ας πούμε, να μην μείνει και να αναρωτιέται τι έγινε τελικά με την καταγγελία του, να ξέρει και τι επιπλοκές μπορεί να έχει αυτό για τον ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα αυτό και κάποια από τα σημεία για το θέμα των αρχών είναι σημεία που όντω μας ενδιαφέρουν και εμάς. Θα δούμε και τις προτάσεις που θα υποβάλουν σχετικά οι άλλες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ. Thank you. I see Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος από το FDD, το ENF, ούτε. Κύριε Σας ευχαριστώ και πάλι. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε η κυρία Τόμ και να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Τόμ ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί ε, και να βρούμε μια σωστή ισορροπία και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κάποιες ε, νομικές ε, ασφαλιστικές ε, δικλείδες ώστε να μην δώσουμε κίνητρα για δυσφημιστικές ή συκοφατικές καταγγελίες. Και πάντοτε εκφράζαμε τη θέση ότι ο φορέας ή το άτομο που είναι το αντικείμενο της καταγγελίας ε, έχουν ε, τεκμήριο θωότητας και φυσικά δικαίωμα υπεράσπισης της θέσης τους. Θεωρούμε ότι η προστασία θα πρέπει να εξαρτάται από την ακρίβεια των πληροφοριών του καταγγέλλοντος. Δεν θα μπορεί ο καθένας να γίνεται καταγγέλλον ε, απλώς κάνοντας κάποιες προσβλητικές ή συκοφαντικές καταγγελίες. Δεν θα πρέπει όλοι άκρητα να τη χάνουν προστασίας. Θα πρέπει να προβλέψουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που μας είπε η κυρία Τόμ ότι θα πρέπει με πολύ ε, προσοχή να το προσεγγίσουμε. Αλλά γι' αυτό και θα συνεχιστούν οι συζητήσεις ε, ώστε ακριβώς να διαμορφώσουμε μια θέση που θα βρίσκεται τη σωστή ισορροπία. Ευχαριστώ. Thank you all for your interview. Εγώ ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Προθεσμία για τις τροπολογίες για αυτή την έκθεση είναι η 18η Ιουλίου, μεσημέρι. Μελέτη των, συζήτηση των τροπολογιών θα γίνει 29-30 Αυγούστου, ψηφοφορία στην Επιτροπή εδώ, στις 24 Σεπτεμβρίου και ψήφο στην Επιτροπή Γιούρι 10 Οκτωβρίου. Προχωρούμε. Στο σημείο 12 τη ημερήσια διάταξη. Γενικός Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, όλα τα τμήματα. Σύντομη παρουσίαση εισαγωγή από εμένα ως Προεδρεύουσας. Υιοθετήσαμε στις 19 ε, Ιουνίου την γνωμοδότησή μας και την εντολή για τον τριμερή διάλογο, δίνοντας τι κατευθυντήρες για τι διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό στην ε, διαπραγματευτική ομάδα. Στο σχέδιο γνωμοδότησή ε, μου τονίζω τι ε, προτεραιότητε της Επιτροπής Απασχόληση, οι γραμμές του προπολογισμού που υποστηρίζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο και τα μέτρα για τους κοινωνικούς εταίρους που αποτελούν την προτεραιότητα για μας όταν μιλούμε για την ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμενο, για παράδειγμα, και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Και δυστυχώς υπάρχει μείωση στις αναλήψεις υποχρεώσεων που προτείνει η Κομισιόν σε σχέση με τις, ε, με τις βιομηχανικές σχέσεις και, τις, και τον κοινωνικό διάλογο. Θα υποβληθούν τροπολογίες για να υπάρξει αύξηση της ανάληψης υποχρεώσεων. Η γνωμοδότηση ε, είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε μείωση του δημοσιονομικού προγράμματος για τα γραμμές που ασχολούνται με τα κοινωνικά δικαιώματα και τη συμπερίληψη. Επιμένω επίσης ότι πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των ε, ε, πληρωμών και των υποχρεώσεων για να επιτρέψουμε να φτάσουν το στόχο τους αυτές οι πολιτικές. Και γι' αυτό Μιλούμε για κάποιες ε, μειώσεις ε, που προτείνει η Κομισιόν στον προϋπολογισμό για το 2019 σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018. Και όπως πάντα θα ε, επαγρυπνούμε για να δούμε τη θέση του Συμβουλίου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο προπολογισμό στις γραμμές που βρίσκονται εντός της δικής μας ε, εντολής δεν θα μειωθεί. Η αρχή ε, επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας επίσης είναι πολύ σημαντική. Η θέση μας ως προς αυτό είναι σαφή. Δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες και νέες θέσεις με νέα φρέσκα κονδύλια θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις ε, υπόλοιπες υπηρεσίες που υπάρχουν. Τούτων λεχθέντων να ακούσουμε σχόλια, αν υπάρχουν σκιώδεις, ο κύριος Διδιέ είναι εδώ, οπότε σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εισηγήτρια. Φτάνουμε σε μία νέα φάση της έκθεσης αυτής με τις τροπολογίες για τον προϋπολογισμό και θέλω να σας ευχαριστήσω. Είχαμε πολύ επικοδομητικές ε, ανταλλαγές απόψεων μέχρι τώρα και μάλιστα και πριν από λίγες ώρες. Συνεργαζόμαστε νομίζω με σωστό τρόπο. Από την αρχή η ομάδα μας, ε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, προσπάθησε να υπογραμμίσει στοιχεία τα οποία θεωρούμε κομβικά στην έκθεσή μας και που περιλαμβάνομαι στην έκθεση την οποία υιοθετήσαμε στις 19 Ιουνίου, δηλαδή απόρριψη κάθε μείωση του προϋπολογισμού, προτεραιότητα στην καταπολέμηση της, τη μακροπρόθεσμη καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ε, ένδυα μια χρήση ορθολογικότερη των διαφθρωτικών μέσων έτσι ώστε αυτή η σημαντικότατη πολιτική να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Και μια πρωτοβουλία για την απασχόληση για τους νέους τις οποίες οι πιστώσεις υποχρεώσεων το 19 δεν πρέπει να μειωθούν σε σχέση με το 2018, δηλαδή 350 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν όμως ορισμένα στοιχεία τα οποία χρήζουν βελτιώσεων. Έχω την αίσθηση ότι θα ήταν σωστό να αναγνωρίσει κανείς από τη μία την μικρή βέβαια αύξηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του τμήματος του σχετικού με την κοινωνική και εδαφική συνοχή. Αυτό ανταποκρίνεται σε σχέση με αυτά τα οποία κάνουμε εμείς στην Επιτροπή μας. Δεύτερον, εκφράζω τη λύπη μου για την μείωση του προγράμματος Κορές κατά 27,5%. Όπως επίσης και του προγράμματος για την μακροοικονομική ε, μακροχρηματοδότηση κατά 28%. Είμαστε αντίθετοι και ελπίζουμε όλα αυτά να περιλαμβάνονται στο κείμενο μετά από την κατάθεση των τροπολογιών. Θεωρώ ότι τα προγράμματα αυτά, τα οποία ασχολούνται με την χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, θα πρέπει τουλάχιστον να μείνουν στο ίδιο ακριβώ επίπεδο το 19 με το 18. Και σχετικά τώρα με τα πιλωτικά προγράμματα, λυπάμαι που η ε, προαξιολόγηση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ακολούθησε τη σωστή κατεύθυνση και αναφέρομαι εδώ στο πιλωτικό πρόγραμμα της κυρίας Κούν για τον μεταστατικό καρκίνο και τον χώρο εργασίας. Έχω την αίσθηση ότι η προσπάθεια ανάλυσης την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν στο ύψος των προσπαθειών τις οποίες έκανε η συνάδελφος και θα θελήσουμε να γίνει μια νέα αξιολόγηση αν και δεν ξέρουμε αν έχουμε πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Και τέλος ενθαρρύνω και καλό από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή να συμπεριλάβει τα στοιχεία για τα οποία πήρε το βαθμό Β ή Α και στον προϋπολογισμό του 19. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα χρησιμοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν γιατί τα πιλωτικά προγράμματα μπορούν να καινοτομήσουν στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα και υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουμε με ταχύτητα γιατί είναι πραγματικές οι ανάγκες οι κοινωνικές που έχουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γιονγκέριος από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Εκπροσωπώ το Σέργιο Πρέιτο, τον σκιώδη συγγετή μας. Εν είδης αγωγής θα ήθελα να πω ότι είναι σαφές ότι ε, είμαστε υπέρ του σχεδίου γνωμοδότησης ε, της εισηγήτριας. Γιατί η Μαρίτα κατάφερε να συμπεριλάβει τις βασικές μας προτεραιότητες το κείμενο, αλλά ξέρεις πώς είμαστε. Θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε παρόλα αυτά την ε, γνωμοδότησή σου και να τη συμπληρώσουμε. Γενικώ χαίρομαι που αναφέρονται οι στόχοι του κοινωνικού πυλώνα, του, ε, των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας του ΟΗΕ. Αυτές είναι πολύ καλές προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2019. Επίσης, ε, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη συνεχώς προσθέτουν νέες προτεραιότητες ε, στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις, επιδεικνύοντας ένα τυφλό εγωισμό, δεν φροντίζουν να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους για να χρηματοδοτηθούν οι κοινέ ευρωπαϊκές πολιτικές και κάτι τέτοιο παρεμποδίζει ε, την αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική ε, ώστε να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες των συμπολιτών μας. Ο συνδυασμό αυτών των δύο ανεύθυνων, κατά τη γνώμη μου, προσεγγίσεων πολύ πιθανό να αυξήσει την απαγοήτευση, την καχυποψία, τη δυσπιστή και τη ματέωση που νιώθουν πολλές φορές οι συμπολίτες μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη γνώμη μας, το κλειδί για τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς για την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα είναι να δημιουργήσουμε συνέργειες ώστε να καταφέρουμε να μειώσουμε τις κοινωνικές διαφορές και ανισότητες που με την παρουσίαση ε, των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ανισότητες και οι διαφορές. Και σίγουρα ε, η περικοπή των προγραμμάτων απασχόλησης κοινωνικών υποθέσεων ε, σε βασικούς τομείς όχι μόνο δεν θα επιλύσει προβλήματα, αλλά θα δημιουργήσει νέα προβλήματα. Ενώ το πρόβλημα της ανισότητας ήδη έχει διαγνωστεί ως το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να αναφέρω τέσσερα προγράμματα. Καταρχήν στην εντολή του προπολογισμού και χάρη στη δική μας πίεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για σημαντικό μηχανισμό που αφορά το μέλλον των νέων, την απασχόληση των νέων, είτε κατοικούν σε αστικά κέντρα, είτε σε στην Ήπεθρο. Πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων ε, και προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα προσωρινά ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τη μακροπρόθεσμη ανισότητα ε, αφιερώνοντας κονδύλια στις ε, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ό,τι αφορά την εγγύηση για τα παιδιά, αντίστοιχο με την εγγύηση για τους νέους, βάζουμε τα παιδιά ως προτεραιότητα και με πρώτα σε αυτό. Θα πρέπει να διορθώσουμε, να εξαλείψουμε την παιδική φτώχεια. Αυτό είναι σημαντική πολιτική προτεραιότητα και θα πρέπει να α, επικεντρωθούμε σε αυτό, αλλιώ θα αποκλείσουμε ένα μεγάλο τμήμα της επόμενης γενιάς. Θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στην προώθηση των ευκαιριών για τι επερχόμενε γενναίε με μηχανισμού που θα εγγυώνται την τα εφόδια σε όλους και τις απαραίτητες υπηρεσίες για να ε, προκόψουν και να γίνουν υπεύθυνα μέλη της κοινωνίας. Και φυσικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την καταπολέμηση της φτώχειας, ιδιαίτερα την εξάλληψη της παιδικής φτώχειας. Και αυτό θα το καταφέρουμε μόνο χάρη στην εφαρμογή μακροπρόθεσμων κοινωνικών δικτών η εγγύηση για τα παιδιά είναι σημαντική διαρθρωτική μεταρρυθμίση και θα πρέπει να θεωρηθεί ως ε, επένδυση στην σταθερότητα και την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που είναι απαραίτητο για την ε, προάσπιση του αναπτυξιακού μας δυναμικού. Επόμενο σημαντικό θέμα, ο κοινωνικός διάλογος. Δεν μπορούμε να ε, στιγματίζουμε, να μιλούμε για αύξηση των μισθών και πιο αξιοπρεπή συνθήκες εργασίας αν δεν ε, ενισχύσουμε τα συνδικάτα και τις οργανώσεις εργαζομένων. Αυτές θα προωθήσουν τη ποιοτική εργασία μέσω στη αμοιβή. Και επίσης, τελευταίο θέμα, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Επιμένουμε γι' αυτό ε, ότι οι νέες πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εις βάρος ε, υφισταμένων και αποτελεσματικών προγραμμάτων. Δεν συμφωνούμε με την έκβαση του τριμερούς διαλόγου, γιατί δεν υπάρχει πια σαφήνεια για τις πηγές χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας αυτής του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και γι' αυτό θα πρέπει στην γνωμοδότησή μας να πούμε με σαφήνεια την άποψή μας. Ευχαριστώ. Κύριε Τρεμπέζος, έχει το λόγο από το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Γενικός Προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 περιλαμβάνει 166 ε, δις ευρώ σε υποχρεώσεις πληρωμών, άρα μιλούμε για αύξηση 3%. Πολλά λεφτά. Και δεδομένου και του Brexit και των ε, εμπορικών διαμαχών που υπάρχουν, εξακολουθούν να είναι αρκετά. Ο προπολογισμό για τις ε, επενδύσεις είναι σημαντικός. Η ιδέα αυτή δεν είναι κακή, αλλά βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχουν αρκετέ αγκυλώσει. Ο προπολογισμό θα πρέπει πάντα να φροντίζει να λύνει τα προβλήματα του ευρωσυστήματο. Άρα εδώ δεν μιλούμε μόνο για το ότι θα πρέπει τα λεφτά να πηγαίνουν στις σωστέ περιφέρειες, αλλά θα πρέπει η να, να, να, χρησιμοποιούνται και σωστά. Μιλούμε για μεταφορές ε, χρημάτων σε πιο φτωχές περιοχές, αλλά αυτό δεν ελέγχεται επαρκώς για τη χρήση και για την ε, δαπάνη τους. Οπότε πρέπει κάπως να μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Ε, η προσέγγιση που προεκτείνεται δεν είναι σωστή. Χρειάζεται περισσότερος έλεγχος, χρειαζόμαστε ανάληψη ευθύνης και χρειαζόταν και πειθαρχία δημοσιονομική. Επίσης, η οι διάφορες δομές ε, που θέλει να προωθήσει η Κομισιόν σύμφωνα με το γαλλικό μοντέλο. Δεν είναι σωστό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατη πρέπει να έχουν τι σωστέ πληροφορίες ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την γραφειοκρατία και την υπερρύθμιση για να μπορέσουν να βοηθήσουν όντως τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ευκαιρίες και για τη βιομηχανία και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασία, γιατί δεν δημιουργούν οι πολιτικές ε, θέσει εργασία. η αγορά το κάνει αυτό. Επίσης, τα κοινωνικά δικαιώματα είναι, είναι πολιτική δήλωση προθέσεων, τίποτε άλλο, δεν είναι κάτι νομοθετικό και το κάνουμε σαν να είναι κάτι παραπάνω τελικά από μια απλή δήλωση προθέσεων. Χρησιμοποιείται ως βάση αυτό για να δικαιολογηθεί η χρήση υπέρογκων ποσών. Δεν θέλω βέβαια να παραπονιάμαι μόνο, θέλω να κάνω και κάποια θετικά σχόλια. Ο προπολογισμό αυτό ενισχύει την προστασία των συνόρων, ε, ενισχύει τα κοινωνικά μα συστήματα και σωστό είναι να υπάρξουν περισσότερα κονδύλια για, την, για τους ε, πρόσφυγες ε, που βρίσκονται στην Τουρκία και για να επανέλθω στην εισαγωγή μου, η τρέχουσα κατάσταση είναι αρκετά καλή προ το παρόν, θα μπορούσε όμω να υπάρξουν και χειρότεροι καιροί, οπότε πρέπει να εξετάσουμε πώ μπορούμε να εφαρμόσουμε και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτά τα περιορισμένα κονδύλια. Ο έλεγχο και τα διάφορα προγράμματα είναι απαραίτητα. Μιλήσαμε πριν για την πρωτοβουλία για του νέου. Εδώ και τέσσερα χρόνια λέμε και ναι, προειδοποιούμε συνέχεια ότι τα αποτελέσματα τη πρωτοβουλία για του νέου πρέπει να ελεγχθούν για να δούμε αν όντω τα, τα κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν σκόπιμα. Πάντα το λέμε και πάντα μας απορρίπτεται το αίτημα. Οπότε πρέπει να δούμε αν όντως τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων ε, δαπανώνται σωστά. Ό,τι και αν κάνουμε, εν ο στόχο της σύγκληση θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Η σύγκληση στην Ευρωζώνη είναι πραγματικά ε, ελλειπής και πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για να τα, να τα μεταφέρουμε στις πιο ε, φτωχές περιοχές. Πρέπει να προσπαθήσουμε με ε, επικοδομητικές λύσεις να υποστηρίξουμε τη δουλειά που έχει να κάνει ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Lamberts. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Υποστηρίζουμε η γενική κατεύθυνση της πρότασής σας. Σχετικά τώρα με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Για μας πάντα αυτό ήταν πάρα πολύ ε, θετικό και η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου λέει ότι αν πρέπει να πετύχει τους στόχους που έχει απαιτεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν να φανούμε προσεκτικοί και να δούμε με ποιο σωστό τρόπο μπορούν να δαπανηθούν οι πιστώσεις αυτές. θα πρέπει να δούμε γιατί υπάρχουν αντιστάσεις στο να ακολουθηθεί αυτή η γραμμή. Νομίζω πάντως ότι είναι πολύ σημαντικό να μην μειώσουμε τα χρήματα τα οποία δαπανούμε στον τομέα τον κοινωνικό. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη. Πάντα μας ζητάνε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο φυσικά και υπάρχουν όρια σε αυτό. Θέλουμε λοιπόν να καταθέσουμε τροπολογίες ενισχύοντας την πρωτοβουλία για τους νέους με λίγα λόγια. Ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι αύριο 12 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει την 29η Αυγούστου το πρωί. Η υποθεσμία για την κατάθεση από πλευράς μεμονωμένων μελών στην Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών η υποθεσμία αυτή δηλαδή όλων αυτών των ομάδων είναι η 6η Σεπτεμβρίου. Κάνουμε προτάσεις λοιπόν για την αναδιανομή των χρημάτων τα οποία ήδη έχουμε, αλλά και για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να βρούμε νέες πηγές χρηματοδότησης. Δεν έχουμε μείνει πολύ, αλλά νομίζω ότι ήταν μια σύντομη και συζήτηση συζήτηση, ε, σύντομη συζήτηση, συγγνώμη. Ε, φτάνουμε στο σημείο 12, ή μάλλον αφήνουμε το 12 και πηγαίνουμε στο 13, ο ρόλος ε, των ε, εργαζομένων στην δημιουργία θέσεων εργασίας για την απορρόφηση της ανεργίας. Η κυρία Βέμπερ έχει το λόγο. Όπως ενθυμίστε συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της πρώτης ανταλλαγής απόψεων, εκφράστηκαν αντίστοιχες απόψεις από όλες τις πολιτικές ομάδες και υπήρξε στήριξη για τη συγκεκριμένη έκθεση. Κατετέθησαν 110 συνολικά τροπολογίες. Από τις τροπολογίες αυτές ε, οδηγηθήκαμε σε 26 συμβιβαστικές. Χθε έγινε μια συνάντηση σε επίπεδο προσωπικού και νομίζω ότι πάρα πολλά θέματα συμφωνήθηκαν ουσιαστικά. Έχουμε στις 28 Αυγούστου μία συνάντηση σκιωδών όπου θα συζητήσουμε και τις συμβιβαστικές. Όπως είπα από την αρχή, η βασική ιδέα δεν είναι να υπάρξουν ρυθμίσεις νομοθετικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων, αλλά να προσπαθήσουμε να επωφεληθούμε τις ε, πρακτικές εμπειρίες, τις χρηστές πρακτικές που υπάρχουν στις διάφορες χώρες, να ανταλλάξουμε κατευθυντήριες γραμμές και εμπειρίες γενικότερα. Και πράγματι υπάρχουν και ορισμένα θέματα τα οποία θα πρέπει να τύχουν προσοχής από πλευράς μας. Ένα από τα θέματα αυτά, ένα από τα πιο σημαντικά, είναι ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται με τέτοιο τρόπο, να καταρτίζονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να κατανοούν σωστά τι σημαίνει αυτή η οικονομική συμμετοχή. Γιατί είναι προφανές ε, ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι που να συνδέονται με αυτή τη δραστηριότητα. Είναι λοιπόν απολύτως φυσικό να κατανοήσουν οι εργαζόμενοι όλα τα συν και τα πλήν αυτής της ε, ρύθμισης. Αυτό μπορεί να γίνει από τις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και από τις υπηρεσίες των κρατών μελών που θα πρέπει να προσπαθήσουν να εξηγήσουν με κατάλληλο τρόπο τις δυνατότητες αυτές. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, κανένας αποκλεισμός, διακρίσεις, θα πρέπει να επιτρέπεται η συμμετοχή όλων των εργαζομένων και επίσης μια σημαντική πλευρά άπτεται του πόσον τι επίπεδο πληροφόρησης μπορούμε να μοιραζόμαστε με τους ενδιαφερομένους Φυσικά δεν μπορούν όλα να δημοσιοποιούνται, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να αποφύγουμε τις καταχρήσεις. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω και θα ακούσω τους συναδέλφους αν τυχόν έχουν ε, κάποιες, ε, κάποιες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα. Κυρία Γιονγκέρος, που ανεκαθιστά το σκιώδηση γιατί του των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Sorry. It's, it's Η κούραση της ημέρας Α, και το πρωί το ίδιο ήταν. κάποιο ξέχασε την κάρτα ψηφοφορίας. Άλλο θέμα αυτό όμω. Εκπροσωπώ τον Εμίλια Πάβελ εδώ που μου ζήτησε, ε, μου ζήτησε να σας διαβιβάσω ότι λείπει που δεν μπορεί να είναι παρόν στις συζητήσεις αλλά μου έδωσε τα σχόλιά του για να το διαβάσω. Σε ό,τι αφορά την θέση του σκιωδού εισηγητού μας θεωρεί ότι η οικονομική συμμετοχή των ε, εργαζομένων μπορεί να αποφέρει καρπούς και ωφέλη και για τους εργαζόμενους και για την επιχείρηση, εφόσον όμως οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στη διαβούλευση, στη λήψη αποφάσεων και αν τέτοια συστήματα συνοδεύονται από κατάλληλη ενημέρωση και κατάρτιση. Σε ό,τι αφορά τα ωφέλη από την πρόταση αυτή, ε, ένα όφελος είναι η βιώσιμη διακυβέρνηση, ο επικοδομητικός κοινωνικός διάλογος και άλλα θέματα όπως η ικανοποίηση των εργαζομένων από την δουλειά τους, ε, η παροχή κινήτρων, οι δυνατότητες ε, ε, αυτοεκπλήρωσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι μόνο αύξηση παραγωγικότητας και της κερδοφορίας. Όπως είπε και η συγγήτρια, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι πλήρως κατατοπισμένοι και ενημερωμένοι γιατί και εδώ υπάρχει κίνδυνος από μια πλημέλη πληροφόρηση. Υπάρχει κίνδυνος α, λόγω του συστήματος αυτού να χάσει ο εργαζόμενος όλη την επένδυσή του ή ακόμη και την δουλειά του αν χρεοκοπήσει η εταιρεία του. Οπότε εδώ θα έχουμε μια διπλή οικονομική ζημία. Εμείς θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων και τα ωφέλη αυτής θα πρέπει να συμπληρώνουν την ε, αμοιβή του που προκύπτει από τη σύμβαση, το δικαίωμα και τις φορές του για την κοινωνική ασφάλεια και να μην υποκαθιστά αυτή η οικονομική συμμετοχή ε, ή να μειώνει την αμοιβή του ή την κοινωνική του εισφορά. Επίσης, ο Μίριαν Πάβελ θα ήθελα να τονίσει ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να γίνεται σε θελοντική βάση για τους ε, ε, Εργαζομένος και να μην επηρεάζει την κινητικότητά τους ή το δικαίωμά τους να ασκήσουν συλλογικές δράσεις. Εν ο σκιώδης ηγητής μας προσβλέπει σε στενή συνεργασία με την εισηγήτρια την κυρία Βέμπερ και τους λοιπούς σκιώδης ηγητές για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ για το έργο σας και περιμένουμε την επόμενη συνάντηση. Ευχαριστώ. Κυρία Σάντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έφτασα κάπως καθυστερημένα γιατί συμμετείχα σε ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ και συζητάτε νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα το σημείο αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάντως την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσή τη. που είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο και αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τη συζήτηση στη βαρύ και μάλιστα βαίνει και προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με τις προτεραιότητες που έχει η ομάδα μας για την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων. Εδώ εξετάζουμε τις 111 τροπολογίες που υπέβαλαν οι συνάδελφοι και εγώ ως σκιώδη συγγήτρια του ΕΛΚ θα ήθελα να υπενθυμίσω τα τρία βασικά μηνύματα που θα θέλαμε να περάσουμε με τις 20 τροπολογίες που καταθέσαμε. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι σίγουρα η οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων των μισθωτών θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να αναπτυχθεί, γιατί αποτελεί ένα τρόπο πιο ακριβοδίκης κατανομής της αξίας στην επιχείρηση. Και θα πρέπει να είναι σε καλό επίπεδο σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει επίσης να σεβαστούμε τα υπάρχοντα συστήματα, καθεστώτα και τις ιδιαιτερότητες των εθνικών ε, επιχειρηματικών ιστών. Σε ευρωπαϊκό πάντως επίπεδο αυτό που θα πρέπει να δημιουργήσουμε είναι ένα χώρο ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών και να δούμε ποια είναι τα εμπόδια στην οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση. Η δεύτερη μας προτεραιότητα είναι η ενισχυμένη οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων να συμβαδίζει με ένα υψηλό επίπεδο ενημέρωσής τους. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να μπορούν να, ε, να διαμορφώσουν εμπεριστατωμένη γνώμη και να αξιολογήσουν σωστά ε, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ενδεχόμενου κινδύνου ε, μια πιθανή οικονομική συμμετοχή του. Επίση, θα πρέπει η οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων να παραμείνει σε εθελοντική βάση και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην ε, είναι δυσανάλογο το κόστος ε, εφαρμογής του συστήματος σε σχέση με τα πιθανά ωφέλη ε, μια τέτοια οικονομική συμμετοχή ή προσφορά στι δυνατότητε οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων του. Πάντω, Χαίρομαι ε, γιατί ε, με ενδιαφέρει πολύ η έκθεση. Ήδη είχαμε μια τεχνική συνάντηση στην οποία πριτάνευσε ένα πολύ θετικό κλίμα και πνεύμα και ελπίζω το ίδιο κλίμα να επικρατήσει και στις επόμενες μας συναντήσεις. Ευχαριστώ κύριο Γκέρικε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Συγγετρία Φέμπερ. Η συμμετοχή των εργαζομένων μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για την κινητοποίηση των εργαζομένων και για την σύνδεσή τους με την επιχείρηση. Ε, ίσως να είναι και ένα στίχημα για τη δική τους την απόδοση μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο, μια νέα κουλτούρα για, την, για το ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να δώσουν τις ιδέες τους και τις πρωτοβουλίες τους στην επιχείρηση. Μπορεί να ενισχύσει το πνεύμα της επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικότητας και χρειάζεται φυσικά για αυτό να υπάρχουν σαφείς κανόνες. Αυτό κάνουμε νομίζω με την συγκεκριμένη έκθεση. Δεν γίνεται οι ε, συγμένε ε, στο χρηματιστήριο επιχειρήσει να υποχρεώνουν την, ε, τη συμμετοχή. Θα πρέπει να απλουστεύσουμε τους κανόνες ώστε στο τέλος να, μπορεί να, ε, να μπορούν να αποφεληθούν όλοι και οι μεσαίες επιχειρήσεις, οι οικογενειακές επιχειρήσεις που θα μπορούν να ενισχύσουν για να δώσουν κίνητρα για τη συμμετοχή των εργαζομένων. Τα κίνητρα αυτά θα θέλαμε να υπάρχουν και όταν θα συζητήσουμε την έκθεση θα πρέπει να εγγυηθούμε την ε, λιγότερη γραφειοκρατία, να εγγυηθούμε προστιθέμενη αξία για τους εργαζόμενους και ε, μείωση της εκμετάλλευσης. Όλα αυτά θα πρέπει να μπουν στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν από κοινού να δημιουργήσουμε μια νέα κουλτούρα ευρωπαϊκή για τη συμμετοχή των ε, Ευρωπαίων, για τη συμμετοχή των εργαζομένων που θα ενισχύσει και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Λάμπερτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που λένε οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι ε, όντως η, ε, το εργασιακό κλίμα είναι ένα σημείο στο οποίο όντως θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ την εισηγητρία για αυτό. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπαν οι οι συνάδελφοι για το ότι όντως τέτοια προγράμματα δεν υπάρχουν για να αντικαταστήσουν ε, τον μισθό. Αυτό είναι θεμελιώδου σημασία, ούτε να αλλάξουν το, κίνδυνο, κυρίω για τα άτομα που δεν είναι σε θέση να αναλάβουν τέτοιου είδου κίνδυνο, αλλά παρόλα αυτά η ενίσχυση και η συμμετοχή των εργαζομένων μπορεί να κινητοποιήσει περισσότερο το εργαδυναμικό δυναμικό. Γιατί σκέφτεται κανείς ότι έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στην εταιρεία για την οποία δουλεύει. Αυτό είναι σημαντικό και βεβαίως το αποτέλεσμα παρόλο που μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερο μοίρασμα του κινδύνου, μπορεί νομίζω να έχει θετικά αποτελέσματα. Κυρίω ό,τι αφορά τι ε, δομέ τι οποίε μελετούμε. Ε, αυτά είναι από τα βασικά σημεία για την εθελοντική φύση που δεν αντικαθιστά το μισθό και που δεν αλλάζει το οικονομικό, τον οικονομικό κίνδυνο. Αλλά τούτων λεχθέντων να μην δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι δημιουργείται μια πανάκια που λύνει όλα τα προβλήματα. Ούτω ή άλλω δεν είναι αυτή η αίσθηση που έχουμε. Είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση, είναι κάτι που όντω μπορεί να ενισχύσει την συμμετοχή. Τώρα δεν ξέρω πόσο μπορεί να κινητοποιήσει τους άνεργους όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι θα βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε, γιατί ούτως ή άλλως την πρόταση ήδη τη βρίσκουμε ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Βέμπερ, θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλες τις βασικές αρχές τις οποίες αναφερθήκατε ήδη συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση και ήδη εφαρμόζονται στην ε, συμβιβαστική πρόταση, στις τροπολογίες δηλαδή. Προφανώς μιλάμε για εθελοντική βάση Προφανώς ε, μιλάμε για συμπληρωματικά έσοδα εκτός μισθού δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι εργαζόμενοι να θυγούν, να πάθουν βλάβες οικονομικές. Και επίσης ε, θα πρέπει να ενημερώνονται με τον σωστό τρόπο, έτσι ώστε να κατανοήσουν κανονικά τους κινδύνους. Έτσι λειτουργεί κάθε επιχειρηματική προσπάθεια. Έχει και επικίνδυνες δραστηριότητες, πλευρές μάλλον, και δεν θέλουμε ο κόσμος να βρεθεί σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι σήμερα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα σχετικά σε κάθε χώρα. Έχω την αίσθηση όμως ότι εδώ έχουμε μία δυνατότητα η οποία δεν χρησιμοποιείται στο βαθμό που θα έπρεπε θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη, θα έλεγα, σταθερότητα στην αγορά απασχόλησης, γιατί ιδιαίτερα σε ορισμένες καλές οικονομικές περιόδους ε, υπάρχουν ε, δυσκολίες να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις σε επίπεδο εργατικού δυναμικού και φυσικά να δημιουργηθούν και νέες θέσεις απασχόλησης. Σας ευχαριστώ λοιπόν και θα τα ξαναπούμε όταν ε, έχουμε τη συνάντηση των σκιωδών στις 28 Αυγούστου και σας εύχομαι ε, καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. 24 Σεπτεμβρίου θα γίνει η τελική ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια θα πάει τον μήνα Νοέμβριο. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε αύριο μια συνάντηση των συντονιστών στις 9 το πρωί μέχρι τις μισή. Μετά ακολουθεί η κανονική συνεδρίαση που θα ασχοληθεί με το κοινωνικό ταμείο και θα έχουμε δύο ώρες για τη συζήτηση αυτή. Ελπίζω κάποιοι από εσά να είναι παρόντες και παρούσες. Έχει σημασία η συζήτηση αυτή. Θα υπάρξει μια εισαγωγή από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντα υπάρχουν απορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δαπανώνται οι πιστώσεις αυτές. Λοιπόν, προσπαθήστε να είστε παρόντες γιατί μετά ξεκινάνε οι πραγματικές διακοπές.